Καλημέρα κύριε και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και καλώ ήρθατε στην αυτή συνεδρίαση της Υποεπιτροπή μας. Σας ενημερώνω ήδη από τώρα για το ότι ορισμένε γλώσσε δεν μεταφράζονται σήμερα. Τα δανέζικα, τα φιλανδικά, τα λετωνικά. Ε, διότι ξέρετε είναι τα πλήρη μέλη, τα μόνιμα μέλη που έχουν προτεραιότητα για να έχουν μετάφραση στις γλώσσες τους. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από το σημείο 4 τα υπόλοιπα σημεία περνάνε με web stream, βγαίνουν στον αέρα δηλαδή, εκτός από το σημείο 4. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την ε, Σουηδική Προεδρία με τον κύριο Σκογ, τον πρέσβη που είναι εδώ μαζί μας. Έπειτα το θέμα της μη διάδοσης το συζητήσουμε την κυρία Ζανέλα που είναι εκπρόσωπος του κυρίου Σολάνα για το θέμα της μη διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για το Γαλιλαίο. Εποφελούμε από την ευκαιρία αυτή, μια που έχουμε εδώ την Σουηδική Προεδρία της ΕΠΑ, για να σας πω ότι εγώ 8 και 9 Νοεμβρίου θα πάω στη Στοκόλμη για να συμμετάσχω στη διάσκεψη Προέδρων των Επιτροπών Άμυνα των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συνεδρίαση η οποία παραδοσιακά λαμβάνει χώρα υπό κάθε Προεδρία. Στην χώρα η οποία σκεί και την Προεδρία. Εννοείται ότι θα σας ενημερώσω μόλις επιστρέψω για το τι έγινε εκεί. Λοιπόν κύριε Πρέσβη, καλώς ήρθατε. Όντως, ήθιστε κατά τη διάρκεια των εργασιών μας να έχουμε την Προεδρία που έρχεται εδώ να εκφράσει τις προτεραιότητες και να μας μιλήσει για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων που θα έχει να κάνει κυρίως με το πώς εξελίσσονται οι διάφορες αποστολές μας και επίση θα θέλαμε να ακούσουμε και για τα διάφορα άλλα σημεία τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για τη Σουηδική Προεδρία. Μα τα εξήγησε και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ο Υπουργό Μπιλ τον Ιούλιο, τον ακούσαμε. Αλλά, εν πάση θα σα δώσω καλύτερα το λόγο για να έχουμε και αρκετό χρόνο μετά για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την εισαγωγή και για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στην υποεπιτροπή σας. Συγχαρητήρια σε όλους για την εκλογή σας και για το ότι είστε σε αυτή την επιτροπή που κατά την άποψή μου πρέπει να είναι πιο συναρπαστική από όλες τις ε, επιτροπές. Χαίρομαι που μπορώ σήμερα να σας απευθύνω τον λόγο και η φιλοδοξία μας θα είναι της Προεδρίας μας δηλαδή, να προσπαθήσουμε να έχουμε έναν όσο δυνατόν πιο επικοδομητικό διάλογο με το Κοινοβούλιο για ζητήματα ΕΠΑ και ΚΕΠΑ και οπωσδήποτε να σας πληροφορούμε τακτικά. Σήμερα, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας. Είναι ακόμα αρχές της Προεδρίας μας, αλλά οπωσδήποτε θα επανέλθω και στο τέλος της Προεδρίας και τότε θα είναι πιο δύσκολη η παρέμβασή μου γιατί τότε θα πρέπει να σας μιλήσω για το εάν επιτύχαμε στο να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιες προτεραιότητες που έχει θέσει για τον εαυτό της και για τα κράτη-μέλη. Οπότε, θα ήθελα τώρα να πω λίγα λόγια, να ξεκινήσω από τη στρατιωτική πλευρά της ΕΠΑ μετά θα περάσω στις ε, πολιτικές ε, πτυχές, θα κάνω κάποια οριζόντια αν θέλετε σχόλια και μετά θα ξεκινήσω να αναφέρω κάποιες από τις προκλήσεις των αποστολών μας. Πριν από αυτό, να πω πως είναι ένα σημαντικό έτος γιατί έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια της ε, ΕΠΑ. Κάποιοι θα έλεγαν πως είναι μια φοβερή επιτυχία αυτή και πρέπει να το γιορτάσουμε. Άλλοι θα πούν πως ε, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα και, θα... και γνωρίζω πως αμφισβητείται η όλη αυτή η πτυχή της ΕΠΑ. Θα ήθελα εγώ να πω πως εγώ θεωρώ πως ε, είναι αξιοσημείωτη η πρόοδος στο θέμα της ε, ΕΠΑ από όταν πρώτα ετέθη η ιδέα και νομίζω πως ε, η αντίληψη που έχουμε τώρα, που είναι αρκετά ρεαλιστική, είναι ότι όσο και αν το συζητάμε εσωτερικά μεταξύ μας, υπάρχει ζήτηση παγκοσμίω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αποστολές και επιχειρήσεις ανά την Ιφίλιο. Και είναι παγκόσμια ε, η δέσμευση αυτή μέχρι στιγμής, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω πως είμαστε σε μια φάση στην οποία αποφασίσαμε να μην κάνουμε κανέναν εορτασμό παρά το ότι κλείνουν 10 χρόνια, αλλά να εξετάσουμε το πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι ελλείψεις και να δούμε πού πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα για να βελτιωθεί αυτό το μέσο που είναι πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της ε, ΚΕΠΑ και όπως σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να έχει τη δυνατότητα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτές τις αποστολές, να τις βελτιώνει και στο εσωτερικό της Ένωσης υπάρχει απέτηση να είναι αποτελεσματικό αυτό το μέσο, να χρησιμοποιείται εφόσον έχουμε δεσμεύσει κάποια κονδύλια και να χρησιμοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτά ω ε, εισαγωγή για τις προτεραιότητε μα. Τώρα στη στρατιωτική πτυχή υπάρχουν τέσσερα θέματα που αποφασίσαμε να εξετάσουμε. Πρώτα απ' όλα οι ομάδες μάχης της Ευρωπαϊκή Ένωσης, μια έννοια που είναι θετική, αλλά είναι σαφές πως ε, δεν χρησιμοποιούνται, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής και πρέπει να γίνει μια πολιτική συζήτηση για το γιατί δεν χρησιμοποιούνται Ίσως να μην έχει υπάρξει το αίτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω πως είναι σημαντικό για τους Υπουργούς Άμυνας ιδιαίτερα της Ένωσης να συζητήσουν το, το ίδιο αυτό το μέσο πρέπει να γίνει πιο εύχριστο, πιο ευέλικτο. Γνωρίζω πως ο στρατηγός ο Μπεντεζάρ ανέφερε αυτά τα πράγματα στην υποεπιτροπή σας την προηγούμενη εβδομάδα και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνα στο τέλος του μήνα, όπου ελπίζουμε να ξεκινήσει μία συζήτηση για να καταλήξουμε σε μία συνένεση, ότι δηλαδή έχουμε αυτές τις μονάδες μάχης για να χρησιμοποιηθούν. Και βεβαίως αυτό έχει πολλές πτυχές και ευχαριστώ να το συζητήσω μαζί σας ε, στις ε, ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν. Ένας δεύτερος ε, τομέας στον οποίο αποφάσισαμε να δώσουμε έμφαση είναι η θαλάσσια επιτήρηση, που είναι δουλειά οριζόντια σε πολλούς πυλώνες, ε, πολλή δουλειά γίνεται από τα κράτη-μέλη όσον αφορά την παρακολούθηση, την ανείχνευση περιβαλλοντικών καταστροφών, οργανωμένου εγκλήματος, ε, μετανάστευσης. Τώρα έχουμε και την επιχείρηση Αταλάντα που βεβαίως χρειάζεται περαιτέρω δυνατότητες ε, θαλάσσιας επιτήρησης και εκεί πέρα η διαλειτουργικότητα στρατιωτικών και πολιτικών ε, συστημάτων και αναγκών μπορεί να βελτιωθεί. Στόχος μας, φιλοδοξία μας, είναι να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων πτυχών της θαλάσσιας επιτήρησης κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας. Τρίτον, η αμυντική βιομηχανία. Πολλά συζητούνται, υπάρχουν διάφορες πτυχές. Αυτό το οποίο εμείς θα θέλαμε να δούμε, ιδιαίτερα όταν τα οικονομικά είναι περιορισμένα, είναι το ζήτημα της εναρμόνισης και της διαφάνειας στις αμυντικές αγορές. Ορισμένε φορές μιλάμε για ανταγωνισμό επίσης όρης, αλλά συγκεκριμένη αυτή η πτυχή είναι εκτός της εσωτερικής αγοράς, αλλά θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρξει ε, μεγαλύτερη διαφάνεια και το πώς γίνονται οι δημόσιες προμήθειες και η αναρμόνιση είναι κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον για να βελτιώσουμε τις ε, διαδικασίες. Γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά στην Κομισιόν, αλλά όπως σας είπα, η Υπουργή Άμυνας καλό θα έκανα να εξετάσουν τον, τον ρόλο τους εδώ. Τέλος, και αυτό νομίζω ταιριάζει και με την γενικότερη τάση να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και την ΕΠΑ, είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη σχέση μεταξύ της Ένωσης και των λοιπόν οργανισμών του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένου ένα πολύπλοκο θέμα. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει πλήρης ε, συνεργασία και λόγοι που είναι πέραν ε, των δυνατοτήτων ε, ενός ψηφίσματος. Δεν μπορώ να αυτό ένα μια απόφαση βεβαίω στου τέσσερι μήνε που απομένουν, αλλά πέραν από τα πολιτικά εμπόδια υπάρχει λόγο να αναζητούμε τρόπου συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Συνεργαζόμαστε σε πολλά θέατρα επιχειρήσεων, Κοσφοπέδιο, Αφγανιστάν και τώρα στην ε, λεκάνη της ε, Σομαλίας και πρέπει από πρακτική πλευρά να δούμε πώς τα πράγματα πηγαίνουν ομαλά. Είναι και θέμα ασφάλειας αλλά και καλύτερης χρήσης των πόρων. Αυτά νομίζω είναι τα τέσσερα θέματα που θα ήθελα να φέρω από τη στρατιωτική πτυχή. Στην πολιτική πτυχή τώρα. Οι απαιτήσει για πολιτικές επιχειρήσεις ΕΠΑ αυξάνονται πάρα πολύ. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Αποτελεί πάγια σουηδική θέση. Εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πολιτικές της δυνατότητες, τις μη στρατιωτικές γιατί όπως σας είπα η ΕΠΑ βεβαίως ε, ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία μας ζητάνε και η προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ότι είναι μια λέσχη προχωρημένων κρατών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και μπορούμε να το εξαγάγουμε αυτό μέσω, της, μέσω των αποστολών μας ε, ανά τον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο θα προσδώσουμε μια παραπάνω αξία. Τι κάναμε λοιπόν, βασιστήκαμε στο έργο των προηγούμενων προεδριών, σε αυτά τα οποία έχει κάνει η γραμματεία της Κομισιόν. Κάναμε μια απογραφή αν θέλετε και να δούμε το τι πρέπει να βελτιωθεί, να μπορούν να γίνουν γρήγορα, να κινητοποιηθούν γρήγορα οι αποστολές, να έχουν τον εξοπλισμό τους και να βρίσκουμε και το κατάλληλο προσωπικό. Αυτό στην ε, μη στρατιωτική πλευρά βεβαίω είναι κάπω δύσκολο. Είναι ήδη δύσκολο στην στρατιωτική πτυχή, αλλά στην μη στρατιωτική υπάρχει... Στη στρατιωτική πτυχή βεβαίω, ε, βεβαίως ο στρατό δεν χρησιμοποιεί το συχνά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαθέσιμος. Ε, η πολιτική πτυχή είναι πιο δύσκολη γιατί η αστυνομία και οι δικαστές έχουν δουλειά ούτως ή άλλως και δεν θεωρούν τα κράτη-μέλη ότι μπορούν να τους ε, στέλνουν στο εξωτερικό γιατί έχουν κενά στο εσωτερικό. Και το θέμα είναι το τι μπορούμε να κάνουμε. Και όπως σας είπα, έχουμε βρει κάποιους ε, τομείς ε, για να προχωρήσει αυτή η συζήτηση. ένα από τα πράγματα που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι κοιτάμε όλα τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε πω κάποια κράτη-μέλη έχουν μεγάλη δυσκολία στο να δώσουν δικαστέ και αστυνομία, άλλε είναι πιο προχωρημένε. Μπορώ να πω ότι οι σκανδιναβικέ χώρε είναι πιο προχωρημένε ε, και έχουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Νομίζω πω οι σκανδιναβικέ χώρε ε, συνεισφέρουν δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό. Ενώ κάποια μεγαλύτερα κράτη-μέλη είναι κάτω από αυτό το οποίο θα περίμενε κανείς Οπότε αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη, οι υπεύθυνοι για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή σε κάθε χώρα, για να μιλήσουν για τις βέλτιστες πρακτικές. Το τι έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό σε εθνικό επίπεδο και αυτό οργανώνουμε τώρα πιο συστηματικά. Στη μη στρατιωτική πλευρά υπάρχουν λεγόμενες ε, ομάδες ε, πολιτικής ε, απόκρισης. Δεν είναι βεβαίως ε, μονάδες μάχης, είναι ομάδες με εμπειρογνωμοσύνη που μπορούν γρήγορα να αναπτυχθούν σε αποστολές ε, διερευνητικές. Θεωρούν πως υπάρχει αυτό το μέσο, δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ συχνά, για την ακρίβεια πάρα πολύ σπάνια το έχουμε χρησιμοποιήσει και θεωρούν πως θα πρέπει να το ξαναδούμε για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε αυτές τις μονάδες ε, πιο γρήγορα. Ένας άλλος τρόπος ε, για να στείλουμε πολιτικό προσωπικό στις αποστολές είναι να έχουμε συχνότερες συναντήσεις μεταξύ των Υπουργών του Δεύτερου και του Τρίτου Πυλώνα. Δηλαδή οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα συζητήσουν τις πτυχές του ΕΠΑ σε ένα συμβούλιο κάποια στιγμή το φθινόπωρο Βεβαίω, επειδή μιλάμε για την πτυχή τη εξωτερική πολιτική, εμεί το θεωρούμε αυτονόητο, αλλά οι Υπουργοί δικαιοσύνη και Εσωτερικών κοιτάνε το εάν έχουν ανθρώπου διαθέσιμου. Ε, και προσπαθούμε λίγο να περάσουμε το επιχείρημα ότι το να καταπολεμάμε την εγκληματικότητα μέσω μια αστυνομική αποστολή στη Βοσνία και να στέλνουμε εκεί την αστυνομία ε, βοηθάει και την εγκληματικότητα, στο να μειωθεί η εγκληματικότητα στη χώρα μας λόγω της παγκοσμιοποίησης του εγκλήματος και είναι και ένα τρόπο για να πείσουμε του Υπουργού Δικαιοσύνη και Εσωτερικών για την ΕΠΑ. Όλα αυτά για να βελτιωθεί η καταπολέμηση της εγκληματικότητας αλλά και για να βρούμε το σωστό προσωπικό για τις αποστολές. Επίσης ε, υπάρχει μία έννοια, ένα σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρι της αστυνομίας, ε, το οποίο είναι από το 2002. Εμείς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να εξτάσουμε εάν είναι σύγχρονο και εξυπηρετεί τις ε, αποστολές μας που αφορούν το κράτος δικαίου και την οργανωμένη εγκληματικότητα. Δηλαδή θα πρέπει η αστυνομία που στέλνουμε να έχει μια κοινή νοοτροπία, οπότε και εκεί πέρα θέλουμε κάποια πρόοδο του ερχόμενου μήνε. Τώρα για τον εξοπλισμό. Και εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα για να φτάνει γρήγορα επί τόπου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει ο κατάλληλο εξοπλισμό. Και εδώ πέρα θα δούμε την ιδέα της αποθήκευση, Ίσως χρειάζεται κάποιο εξοπλισμό να είναι διαθέσιμος σε κάποιες αποθήκες για να μπορεί να αποστέλλεται γρήγορα μαζί με το προσωπικό εάν χρειάζεται οι αποστολές να φύγουν γρήγορα. Και ένα σχετικό ζήτημα είναι οι προμήθειες. Αποδεικνύεται, όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύπλοκους κανόνες για τις προμήθειες ε, για να διασφαλίσουμε πως ε, αυτός ο οποίος θα κάνει την καλύτερη προσφορά θα πάρει και το συμβόλαιο και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια κτλ. Αλλά αυτό δυστυχώς όταν μιλάμε για γρήγορη ανάπτυξη αποστολών ΕΠΑ σημαίνει προβλήματα γιατί οι καθυστερήσεις για αλεξίσφαιρα γυλαίκα ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό έχουν καθυστερήσει. Και δεν έχει νόημα να στέλνουμε προσωπικό πολίτε στο Αφγανιστάν, α πούμε, χωρίς ε, τον κατάλληλο εξοπλισμό. Οπότε θα δούμε αν μπορεί να υπογράψει η Κομισιόν μια συμφωνία πλαίσιο για να υπάρχει ένας κατάλογος προμηθευτών οι οποίοι εκ των προτέρων θα μπορούν να προμηθεύουν γρήγορα και με αξιοπιστία αυτό το υλικό. Αυτά εν συντομία το τι σκοπεύουμε να κάνουμε στη μη στρατιωτική πλευρά. Υπάρχουν κάποια οριζόντια ζητήματα που αφορούν και τις πολιτικές και τις στρατιωτικές ε, αποστολές. Το ένα είναι η συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής πτυχής. Ένα ζήτημα το οποίο σκοπεύουμε να δούμε από την πτυχή της ε, ανάπτυξης των δυνατοτήτων Ξέρετε πως υπάρχει ένας στόχος ε, και από πλευράς ε, πολιτικής για το 2010 που και από πλευρά στρατιωτική. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να τα συνδυάσουμε, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να υπάρξει κάποια συνέργεια. Και παραδείγματο χάρη, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολιτική αποστολή στη Βοσνία και μια στρατιωτική. Οπότε θεωρούμε το ότι για να εξοικονομήσουμε χρήμα και πόρους. Όσον αφορά την επιμελητία π.χ. μπορεί να είναι αυτή κοινή. Αλλά υπάρχει βεβαίως πάντα και υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και νοοτροπίες. Αλλά είναι ένας τομέας που αξίζει να εξετάσουμε. Επίσης, όπως είπα, θεωρώ πως ένα από τα θετικά της ε, ΕΠΑΑ και εκεί πέρα που είμαστε πιο προχωρημένοι σε σχέση με άλλους οργανισμούς είναι ακριβώς τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, είτε στρατιωτικά είτε πολιτικά. Και αν ε, καταφέρουμε να ρυθμίσουμε αυτό το μείγμα καλύτερα από ό,τι σήμερα ήδη από την φάση του προγραμματισμού θα έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Ένα άλλο θέμα που θεωρούμε ότι έχει μείνει πίσω όσον αφορά τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαιτησία. Στο φάσμα των μέσων που έχει στην διάθεσή της η ΕΠΑ και η ΚΕΠΑ, η διαιτησία κάποιες φορές έχει αποτελε... αποδειχθεί αποτελεσματική Έχουμε τον ε, κύριο Σολάνα που είναι πολύ καλός διαπραγματευτής με αρχηγούς κατών κυβερνήσεων όπως π.χ. στην Ουκρανία με την Πορτοκαλή Επανάσταση. Είχαμε στην ε, Πουγουδουμού πολύ καλή διατησία με τις συμφωνίες της Αχρίδας ε, και υπάρχει, υπάρχουν και οι ειδικοί απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επί καθημερινής βασίως αντιμετωπίζουν δύσκολες συγκρούσεις και θέλαμε να δούμε λίγο το εάν ε, τους στηρίζουμε αρκετά, τους εκπαιδεύουμε αρκετά, αν έχουν αρκετή οργανωτική στήριξη. Για τον λόγο αυτό τους μαζέψαμε όλους σε ένα δωμάτιο τον Ιούλιο και ο κύριος Καλμπίλτ και ο κύριος Σολάνα για να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει αυτές τις δυνατότητες στον τομέα της διατησίας. Οι πτυχές του φίλου. Δεν θα σας εκπλήξει το ότι ακούτε από τη Σουηδική Προεδρία το ότι είναι σημαντικές αυτές οι πτυχές. Έχουμε προωθήσει αυτά τα θέματα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε οπωσδήποτε. Θα δούμε συγκεκριμένα την κατάρτιση έτσι ώστε όσοι αποστέλλονται σε αποστολές ΕΠΑ είναι παρκώς καταρτισμένοι για τις πολιτικές του φίλου και έχουν κώδικες συμπεριφορά όσον αφορά την αντιμετώπιση ορισμένων λεπτών ζητημάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικώ είναι ένας άλλο τομέα. Είπα πριν πω ε, ένας από τους λόγους για τους οποίους μα ζητάνε, εξακολουθούν να ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα ρόλο σε συγκρούσει, είναι το γεγονός πως είμαστε αρκετά αξιόπιστο οργανισμό η Ένωση, όταν μιλάμε για την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό και απαιτείται από εμά να επιδείξουμε γνώση και σεβασμό όταν μιλάμε για εξαγωγή ε, τρόπων την αυτών των αξιών. Και βεβαίως οι αποστολές αυτές της ΕΠΑ δεν είναι κάποια εξαίρεση, πρέπει να είναι το υπόδειγμα του πώς ε, δουλεύουμε. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας, ε, όπου λαμβάνουμε όλο και περισσότερα αιτήματα. Είναι σημαντική πτυχή, πτυχή του τι κάνουμε στο Κόγκο, τη Λαϊκή Δημοκρατία, στη Γουινέα Μπισάου. Οπότε πρέπει να υπάρχει και ανάλογη οργάνωση εντός των κρατών μελών. Το ξεκίνησε αυτό η Γαλλική Προεδρία. Τέλος, όσον αφορά την εξέλιξη της ε, ΕΠΑ. Δεν πρέπει και να χαιρόμαστε πολύ. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Ένας τρόπος ε, ε, διάρκους βελτίωσης βεβαίως είναι η το να διδασκόμαστε από αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Δηλαδή πρέπει να επανεξετάζουμε τις αποστολές μας, να δούμε πότε έχουμε κάνει λάθη, να είμαστε ειλικρινεί ω προ αυτό. Και για να είναι σοβαρή αυτή η διαδικασία πρέπει να είμαστε τελείω ειλικρινεί για το ποια είναι τα μαθήματα που αντλήσαμε. Και ορισμένε φορέ αυτό σημαίνει πω πρέπει να έρθει κάποιο απ' έξω. Δηλαδή κάποιο που αντιλαμβάνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έρχεται απ' έξω για να αξιολογήσει το τι γίνεται. Και εκεί πέρα μπορούμε να βελτιωθούμε. Και αυτό νομίζω είναι προς ε, το συμφέρον το δικό σας. Ε, να υπάρχει διαφάνεια δηλαδή όσον αφορά τη... τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω αναφέροντας κάποιες επιχειρήσεις, δεν θα τις αναφέρω όλες. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτές οι οποίες ε, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να απασχολήσουν την Επιτροπή σας και τη δική μου Επιτροπή, την ΕΠΑ τους ε, ερχόμενους μήνες. Πρώτα απ' όλα στη Βοσνία, όπου βεβαίως ε, έχουμε στρατιωτική ε, αποστολή, όπως ξέρετε, τη U4 Altea και την πολιτική, την αστυνομική αποστολή εδώ και χρόνια. Και είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Η στρατιωτική αποστολή με 2.000 άντρες έχει σχεδόν ολοκληρώσει την εντολή της επιτυχώς και είναι θέμα του να έχουμε τώρα μία μετάπτωση σε μία πολύ πιο μικρή παρουσία που κυρίως στόχο θα έχει την εκπαίδευση. Αυτή η μετάπτωση βεβαίω θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί περισσότερη ένταση στη Βοσνία και θα πρέπει να συντονιστούμε και με το κλείσιμο των γραφείων του είπα του εκπροσώπου Οπότε να γίνει η διαδικασία του Dayton μια διαδικασία των Βρυξελών για να μπορέσει να ενταχθεί και η Βοσνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις απαιτήσει ε, που έχει αυτό. Για να συμβεί βεβαίως κάτι τέτοιο πρέπει να έχει κλείσει το γραφείο του ΙΠΑ του αλλά όπως σας είπα πρέπει να συντονιστεί αυτό με τη στρατιωτική επιχείρηση. Στο κοσφοπέδιο είμαι σίγουρος πως έχετε ενημερωθεί. Νομίζω Πίτερ Φράιτ είχε έρθει εδώ. Α, όχι, στην Επιτροπή Εξωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρετε πως υπάρχει μια συζήτηση για την ανάγκη υπογραφή ενό αστυνομικού πρωτόκολλου με τη Σερβία. Πρέπει να λειτουργήσει η Γιουλέξ και να κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό σε ένα περιβάλλον που έχει περιπλοκές. Απλά θα ήθελα να πω πως το ικανοποιητικό για την EULEX είναι μια τεράστια αποστολή, ε, την υποδέχονται όλοι θετικά, αλλά είναι ε, δύσκολο το περιβάλλον. Πέντε κράτη-μέλη της Ένωσης δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσφοπέδιο, αλλά ε, υποστηρίζουν όλες οι χώρες και οι 27 την αποστολή αυτή και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό τη στιγμή που γίνεται επιχειρησιακή αυτή η αποστολή και καταλήγει να είναι στο, στην πρώτη γραμμή των δύσκολων ζητημάτων που αφορούν ε, την ε, επαφή των διαφόρων αστυνοτικών ομάδων στο κοσμοπέδιο. Το βλέπουμε αυτό ήδη και εμείς σκοπεύουμε να είμαστε στιβαροί όσον αφορά τα συμφέροντα της EU Δηλαδή η Πριστίνα πρέπει να συνεργαστεί με την ε, αποστολή αυτή, η οποία σκοπεύει να υπηρετήσει όλες τις κοινότητες του κοσφοπεδίου. Στο Αφγανιστάν, ένα ζήτημα που συζητάνε οι Υπουργοί και Εξωτερικών και Άμυνας, το ρόλο δηλαδή της Ένωσης, να μην ξεχνάμε και την αστυνομική μας ε, αποστολή, την EUPOL, έχει ληφθεί η απόφαση να αυξηθεί σε 400 άτομα και προσπαθούμε ακόμα να βρούμε τους κατάλληλους αυτούς επαγγελματίες για τις αποστολές αυτές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά αυτό εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη, το πόσο θα, θα συνεισφέρουν, κάτι το οποίο δεν κάνουν σήμερα δυστυχώς. Οπότε πρέπει να μας στηρίξετε και εσείς κάνει πολύ σημαντικό έργο αυτή η αποστολή, κάτι που αναγνωρίζουν και οι ΙΠΑ και οι Αφγανικές Αρχές και ο Υπουργό Εσωτερικών ότι η αστυνομική αποστολή ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα της ε, εκπαίδευσης και της συνεργασίας με την αστυνομία. Μια αξιόπιστη αστυνομία στο Αφγανιστάν είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε τη στρατιωτική μας ε, παρουσία μακροπρόθεσμα. Στη Γεωργία γνωρίζετε πως εκλήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ γρήγορα να αναπτύξει μια αποστολή και το καταφέραμε και προξένηξε έκπληξη. Βεβαίως δεν είχαμε σοβαρά επεισόδια, αλλά είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο και δεν ε, βελτιώθηκε η κατάσταση μετά την ε, αναχώρηση των αποστολών του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ λόγω έλλειψης ε, συνεργασίας και από πλευράς της Ρωσίας. Και εδώ πέρα προσπαθούμε να ορίσουμε τον ρόλο της αποστολής παρατηρητών της Ένωσης δεδομένης και της ε, κατάστασης που έχει διαμορφωθεί ότι δηλαδή οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη παρουσία εκεί πέρα. Η Αταλάντα, η επιχείρηση στα ανοιχτά της ε, Σομαλίας. Είναι νομίζω μια πολύ επιτυχημένη αποστολή. Τα κράτη-μέλη συνεισφέρουν και έρχονται και νέες συνεισφορές. Άπατελεσε απάντηση στο πολύ επίγον ζήτημα της πειρατείας που εμποδίζει και την διεθνή κοινότητα στο να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Σομαλία. Το πρόγραμμα, το επισητιστικό του ΟΗΕ μας είπε πως βοηθήθηκε πάρα πολύ από αυτή την αποστολή, οπότε έτσι βελτιώνεται και η ζωή των Σομαλών. Εμείς θεωρούμε πως αυτό είναι κατοθετικό και πρέπει να συνεχιστεί, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί και με περισσότερες προσπάθειες ε, στην ξηρά στη Σομαλία. Να βελτιώσουμε την μεταβατική κυβέρνηση και βεβαίως να έχουμε κατά νου και το συμφέρον των Σομαλών. Οπότε το Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιούλιο να δει μια σειρά τομέων στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σομαλία για να συμπληρώσει την επιχείρηση αυτή κατά της πειρατείας με κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε πως αυτό είναι πολύ δύσκολο, η κατάσταση λεωρά ασφαλείας είναι δύσκολη, αλλά αυτό γίνεται σε στενό συντονισμό και με τον ΟΗΕ και τη ΣΥΠΑ. Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ, υπάρχουν και άλλες σημαντικές αποστολές, αλλά φαντάζομαι πως θα με ρωτήσετε και όλες για αυτές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω και τις ε, ερωτήσεις σας, αλλά και τις συμβουλές σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη για την παρουσίαση την τόσο πλήρη που μας κάνατε. Σίγουρα οι ερωτήσεις θα είναι πολλές και τα σχόλια μεταξύ των συναδέρφων. Θα ήθελα όμως πριν δώσω το λόγο στους συναδέρφους, να σας ρωτήσω δύο πράγματα για τα οποία θα ήθελα να σας ακούσω να μας λέτε περισσότερα. Τις ομάδες μάχης battle groups. Είναι μια καλή ιδέα που δεν χρησιμοποιείται αρκετά. Γιατί, γιατί δεν λειτουργεί. Πριν την συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας τέλη Σεπτεμβρίου, μήπως έχετε κάποια ιδέα τι θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτή τη διαπίστωση. Και έπειτα για την αποστολή Αταλάντα. Πέρα από την επιτυχία που έχει για να ε, καταπολεμήσει την πειρατεία, έχουμε όντω καλά ε, νούμερα που από διάφορες υπηρεσίες όπως ο ΠΑΜ που εποφελούνται από την δράση αυτή. Έχουμε συμφωνίες και με τις αρχές της Κένιας, γιατί από ό,τι φαίνεται ένα από τα προβλήματα τα οποία συνεχώς εμφανίζονται είναι δικαστικά τι ε, γίνεται στην Κένια όταν συλλαμβάνονται κάποιοι πειρατές. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά το λόγο η συναδελφή μου και πρώτα απ' όλα ο κύριος Φανόρδεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Σκόκ για τα τόσο διαβοτιστικά που μας παρουσίασε για το τι συμβαίνει με την ΕΠΑ και ποιες είναι οι προτεραιότητες σήμερα. Είπατε ότι το να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της ΕΠΑ δεν το κάνουμε επειδή δεν έχει γίνει περισσότερη πρόοδος από όσοι <clears throat> έχει γίνει. Από την άλλη μεριά όμως η ΕΠΑ δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε να ξεκινήσει. Ουσιαστικά δεν έχει γίνει αυτό που θα θέλαμε πραγματικά να γίνει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. ούτε τα θέματα τα οποία χειριζόμαστε και με το ΝΑΤΟ έχουν προχωρήσει όπως θα θέλαμε. Υπάρχει κάποια έμμονη ιδέα με αυτές τις περίφημες ομάδες μάχης, που εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Εμένα, για παράδειγμα, με εκπλήσει που δεν είπατε περισσότερο για το Αφγανιστάν σήμερα. Το Αφγανιστάν, βλέπετε, είναι η κύρια ανησυχία όλων μας. Γιατί αν δεν πάνε καλά τα πράγματα στο Αφγανιστάν, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες. Και όταν λέω να πάνε καλά τα πράγματα, δεν εννοώ να συνεχίσουμε να κυνηγάμε ε, τους στόχους που έχουμε κυνηγήσει τους τελευταίους μήνες και χρόνια, αλλά νομίζω ότι όλοι μας, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ, ακόμα και ουδέτερες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή στο Αφγανιστάν 400 Σουηδοί μάλιστα στην ε, ICF, την αποστολή ICF. Και μάλιστα είχατε και απώλειες. Χαιρετίζω την ε, παρουσία και τη συμμετοχή της Σουηδίας, αλλά γι' αυτό με εκπλήσει το γεγονός ότι η ΕΠΑ δεν επικεντρώνεται στο Αφγανιστάν δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι. Έτσι μόλις αναφερθήκατε εσείς στη Νιούπολ, μα ειλικρινά, είναι καταστροφή από την αρχή. Πάλαμε χρήματα, δαπανήθηκαν πολλά, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Είναι ζωτική σημασία όμως η κατάρτιση ε, της ε, αστυνομίας του Αφγανιστάν είναι αποτελεσματική να αποδώσει. Οι Αμερικανοί επίσης έχουν βάλει πολλά. Γι' αυτό λοιπόν μήπως θα έπρεπε να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει, συντονίζει τις δικές της δραστηριότητες στο Αφγανιστάν. Μπορεί, αλλά σίγουρα όχι και με τον ΝΑΤΟ, ενώ θα μπορούσε. Και αυτή είναι μια άλλη ανησυχία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει επίσης και στο μη στρατιωτικό τομέα. Και έχουν γίνει πολλά στο Αφγανιστάν, στο μη στρατιωτικό τομέα. Ανοικοδόμηση, ανάπτυξη, στους τέσσερις τομείς ε, δύσκολους από πλευράς ε, ασφάλειας. Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα σε στενή συνεργασία όμως με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και άλλοι τομείς για τους οποίους θα ήθελα να ακούσω περισσότερα, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, αλλά να πιστεύω πως τη στιγμή αυτή η προσπάθειά σας πρέπει να είναι το Αφγανιστάν και το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο Αφγανιστάν. Γιατί είναι ζωτική σημασία η περιοχή αυτή για όλους μας. Ευχαριστούμε, κύριο Πασκού. Ευχαριστώ. Ναι. Ίσως μπορούμε βέβαια να συζητήσουμε κατά πόσο καλά ξεκινήσαμε ή όχι με την ΕΠΑ. περιπτώσει τώρα υπάρχει, έχουμε τη συμφωνία που έχουμε, έγινε από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει, ας προσπαθήσουμε να την κάνουμε και να λειτουργήσει. Μπορεί να ακούγεται φιλοσοφικό αυτό που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η φιλοσοφία εφαρμόζουν και οι Σουηδοί και οποιαδήποτε άλλη προεδρία είχαμε για αυτά τα θέματα. Συμφωνώ και μαζί σα για το ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα έπρεπε να διευκρινιστούν. Έχω λοιπόν και εγώ μερικά. Πρώτον, ακόμα και μετά από την παρουσίαση αυτή του πρέσβη, είναι προφηνές ότι ο Ντομινίκ Μωσή είχε δίκιο όταν έλεγε ότι ο Ατλαντικός είναι χωρισμένο στα δύο από το ναι μπορούμε που είναι Αμερική και ναι θα μπορούσαμε που είναι η Ευρώπη. Σωστό. Όσον αφορά τώρα τις ομάδες μάχης, γιατί έχουμε τις ομάδες μάχης ενώ εμείς έχουμε διαφορετικές δυνάμεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εν μέρη γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ομάδες μάχης. Δεν έχει επιτευχθεί συνένεση. Αν μία από τις χώρες που συμμετέχει στις ε, ομάδες μάχης δεν συμφωνεί με την οργάνωσή τους, ε, δεν μπορούν και να χρησιμοποιηθούν. Δεύτερον, ή οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουμε δεν αντιστοιχούν στα καθήκοντα των ομάδων μάχης ή ομάδες μάχης δεν είναι φτιαγμένε έτσι ώστε να είναι καλές για τις επιχειρήσεις που θέλουμε να τι χρησιμοποιήσουμε. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα μια διαφορά πάντως ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις ομάδες μάχης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Έπειτα υπάρχει και κάτι άλλο. Η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία των ομάδων μάχης. Ξέρετε ότι ο εφιάλτης των σχεδιαστών ε, μάχης είναι το να χρησιμοποιούν δυνάμεις που έχουν ε, ετοιμαστεί για κάτι άλλο και να τις χρησιμοποιούμε για τις ομάδες μάχης. Αυτό είναι ο φιάλτης. Και είναι η καλύτερη συνταγή για να ε, χάσουμε κάθε δυνατότητα δράσης. Για να μπλοκάρουμε τα πάντα. Οπότε, πέρα από το πολιτικό σκέλος, που πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό, υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Κάτι άλλο. Έχουμε την επιτήρηση στη θάλασσα, ναι. Έχουμε τη γνώση του τι γίνεται γύρω μας, στα ύδατα. Ναι, αλλά γιατί για να μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, άπαξ και το απαιτούν οι καταστάσεις. Η θαλάσσια επιτήρηση πρέπει λοιπόν να συνδέεται με τη δυνατότητα παρέμβαση, επέμβαση. Τώρα, σε ποιε περιπτώσει αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν πρόκειται για φυσικέ καταστροφέ, θεομηνίε, όταν πρόκειται για παράνομη μετανάστευση ή το να λυθούν κάποια νομικά ζητήματα. Ξέρετε, ωραία, άντε και του πιάσαμε. Και μετά τι θα του κάνουμε, του πειρατέ, α υποθέσουμε. Βλέπετε, όλη την αλυσίδα πρέπει να εξετάσουμε. Δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στα τεχνικά ζήματα που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση στη θάλασσα, αλλά μετά τι κάνουμε, άντε επιτηρήσαμε, άντε βρήκαμε το λάθος, άντε τους πιάσαμε. Μετά πρέπει όλη την αλυσίδα να την εξετάσουμε και να ξέρουμε τι περιλαμβάνει. Έπειτα, για τον εξοπλισμό, βλέπετε η εξωτερική πολιτική κατά ψέματα είναι εθνική πολιτική. ως επιτοπλίστων. Αλλά τώρα αυτά τα μικρά πραγματάκια που αναφέρατε, συμφωνίες, πλαίσιο κτλ. Αυτά μπορούν να γίνουν και θα έπρεπε να συνεχίζονται. Και η διαμεσολάβηση ναι. Θέλουμε, άπαξ και μπορούμε να βοηθήσουμε να είμαστε διαμεσολαβητές. Αλλιώς θα είναι άλλοι αντί για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ. Για να επανέλθω στην φράση του κυρίου Πασκού, για την ώρα για το Αφγανιστάν κανένας δεν λέει yes we can, ναι μπορούμε. Όλοι λένε yes we should, θα μπορούσαμε. Ε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα πρέπει να γίνει. Έχω να κάνω, ωστόσο, κάποιες πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είπατε κύριε Σκόγκ, ότι οι ομάδες μάχης έχουν δημιουργηθεί για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σαν να κατηγορείτε τους προηγούμενους για το ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά τα προηγούμενα χρόνια ή μήνες. Ε, με ενδιαφέρει αν εσείς πιστεύετε ότι σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις στο παρελθόν θα μπορούσαμε να έχουμε χρησιμοποιήσει περισσότερο αυτές τις ομάδες τις μάχημες. Ας πούμε μια αποστολή στο τσάντ ή οπουδήποτε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις δηλαδή και έπειτα για την ε, επιτήρηση την θαλάσσια είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Το να πείσουμε τους πολίτες μας για την αναγκαιότητα μιας ε, κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας είναι ένα από τα παραδείγματα όπου μπορούμε εδώ να δείξουμε, να αποδείξουμε στους πολίτες πόσο σημαντικό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι. Σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις εθνικές προσπάθειες κτλ. Δεν είναι θέμα όμως του ΝΑΤΟ ή, το ή θέμα κάποιας εθνικής κυβέρνησης είναι πραγματικά ευρωπαϊκό ζήτημα. Το θέμα ασφάλειας ε, σε σχέση με την πειρατεία, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Επίσης αναφέρατε, λειτουργεί, πώς λειτουργεί, πού υπάρχουν προβλήματα. Η Προεδρία σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα για να πείσει τους πολίτες πόσο σημαντικό είναι ίσως να μην πείσετε τον κύριο Φανόρντεν, αλλά αν πάση περιπτώσει κάποιος άλλος μπορεί να τους πείσετε για τη σημασία της ε, ευρωπαϊκής κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Γιατί σε αυτό το επίπεδο πραγματικά υπάρχει ε, ένα μείγμα ε, πολιτικής και στρατιωτικής δράσης. Υπάρχουν θέματα περιβαλλοντικά. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λοιπόν πόσο ικανοποιημένο ή όχι είστε με το συντονισμό που γίνεται και τι μπορείτε να κάνετε για να το βελτιώσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ και μετά θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Πρέσβη για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν τόσες πολλές ερωτήσεις για τις ομάδες μάχης που σχεδόν δεν τολμάω να κάνω κι εγώ ερώτηση για το ίδιο πράγμα, αλλά μία σύντομη ερώτηση. Ποια επιχειρήματα κατά της χρησιμοποίησής τους πρέπει να ξεπεράσετε για να χρησιμοποιηθούν τι, τι λέει π.χ. κάποιο κράτος ε, για να φέρει η αντίρρηση. Κατά τα λοιπά, σας ευχαριστώ για την ευρύ παρουσίαση των θεμάτων της ε, Προεδρίας σας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι για την Γιούπολ στο Αφγανιστάν. Ξέρετε πως και οι Αμερικανοί εκπαιδεύουν την αστυνομία και υπήρχαν παράπονα πως έχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις Εν τω μεταξύ έχουμε συμφωνήσει με τους Αμερικάνους ε, για το που στοχεύει η εκπαίδευσή τους ε, των Αφγανών. Και κάτι ακόμα, δεν υπάρχει κάποια ισχυρή κεντρική παράδοση έτσι, κράτους ε, στο Αφγανιστάν. Γιατί εκπαιδεύονται αυτοί οι αστυνομικοί κεντρικά και μετά αποστέλλονται στις επαρχίες. Μήπως υπάρχει ο κίνδυνος εκεί οι ντόπιοι να τους δουν ως ξένο σώμα, να μην πως ξένα στρατεύματα. Μήπως θα έπρεπε αποκεντρωμένα επί τόπου να εκπαιδεύσουμε νομικού ντόπιου που θα δουλέψουν και εκεί που βρίσκονται. Ένα ερώτημα ακόμα. Αμέσως μετά θα δείτε πως ακολουθεί η κυρία Τζιανέλα και έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα μη διάδοσης ε, και την αναθεώρηση της σχετικής συνθήκης. Πού βρισκόμαστε στην προετοιμασία των, ε, των διαπραγματεύσεων αυτών για την ε, συνθήκη μη διάδοσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για τις πρώτες αυτές ερωτήσεις. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σχολιάσω τις ερωτήσεις και βέβαια τις συμβουλές που ε, μου προτείνατε θα έχω όλα σημειώσει. Για τις ομάδες σε μάχη. θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από αυτόν. Έχω την εντύπωση ότι Ίσως υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά την πολιτική δέσμευση εδώ και μιλώ πολύ ανοιχτά σχετικά με την σουηδική εμπειρία. Ήμασταν ε, ένα έθνος πλαίσιο για πέρσι ε, για μία από τις ομάδες μάχης, ε, την βόρεια ομάδα μάχης. Ήταν πολύ μεγάλη επένδυση για μας, πολύ σοβαρή επένδυση. Δεν χρησιμοποιήθηκε διότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες περιστάσεις για να χρησιμοποιηθεί. Εμείς κάναμε αυτή την επένδυση βέβαια με ενδιαφέρον, ε, ενδιαφερόμενοι μάλλον να τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Ε, ίσως να τοποθετούν στοιχεία σε αυτές τις ομάδες μάχης που δεν υπάρχουν πραγματικά, μάλλον που δεν τοποθετούνται πραγματικά για να χρησιμοποιηθούν. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν λέω πως όντως συμβαίνει αυτό, αλλά πιστεύω πως θα ήταν σκόπιμο να συζητηθεί. Υπάρχει το θέμα της χρηματοδότηση, υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό κοινό κόστος όλα αυτά, ακόμα και αν τα ε, στρατεύματα δεν βρίσκονται μέσα στην ίδια την ομάδα μάχης, σημαίνουν κόστος για όλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για ορισμένους μεγάλο κόστος. Ακόμα όπως είπα και αν τα στρατεύματα αυτά δεν βρίσκονται επί τόπου. Μπορεί μάλιστα το κόστος να είναι απαγορευτικό για ορισμένου. Έπειτα, η ιδέα για αυτές τις ομάδες μάχης είναι το να μπορούν να, αναπτυχθούν πολύ γρήγορα και αυτό μπορεί να είναι πραγματικό όταν θέλουμε να δούμε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη, η στρατηγική δηλαδή ε, αερομεταφορά. Και αυτό είναι θέμα και για τον ΝΑΤΟ. Μπορεί να υπάρχουν τα στρατεύματα, αλλά το να μετακινηθούν γρήγορα επί τόπου είναι κάποιες φορές προβληματικό λόγω της έλλειψης στρατηγικών αερομεταφορών. Αυτά είναι λοιπόν ζητήματα που πιστεύουμε πως θα πρέπει να συζητηθούν. Θα πρέπει να είμαστε ίσως πιο ευέλικτοι Ίσως να μην χρειάζεται να μετακινηθεί μια ολόκληρη ομάδα μάχης. Αν υπάρχουν δύο ας πούμε μόνιμες ομάδες μάχης, θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε κάποια κομμάτια για μια άσκηση ας πούμε τέταρτης γενεάς. Ένα παράδειγμα για μια πολύ παρατεταμένη άσκηση τέταρτης γενεάς. Υπήρχαν ομάδες μάχης τότε. Θα μπορούσαμε ίσως να αφαιρέσουμε κάποια τμήματα αυτής της ομάδας μάχης είτε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη στρατηγική, στρατηγικό απόθεμα, αποθεματικό για κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Η εφεδρία ε, μια στρατηγική εφεδρεία να υπάρχει τέτοιο τέτοιου είδους ε, στόχους. Υπάρχει, υπήρχε το θέμα της, ε, του Κονγκό. Στον Ανατολικό Κονγκό η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλοί κόσμος επιτόπου και πραγματικά μια, μια μη ρεαλιστική εικόνα για την καταστροφή που, που συνέβη μάλλον στα τέλη του περασμένου χρόνου. Ορισμένοι εξημών τότε και υπήρχε μια επιστολή από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σκεφτεί μήπως στείλει μια ομάδα μάχη σε εκείνη την φάση και ορισμένοι από εμά θεωρήσαμε ότι έπρεπε να το συζητήσουμε ενώ άλλοι όχι. Ίσως το θέμα να έχει εν μέρη ληφθεί μέσω πολιτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Κισάσα και το Κιγκάλι αργότερα, αλλά βέβαια με τεράστια ανθρωπιστικά προβλήματα. Δεν λέω πω η ομάδα μάχης θα τα χελίσει όλα αυτά, αλλά υπήρξε μια περίπτωση όπου αυτό συζητήθηκε και εκεί νομίζω θεωρήσαμε πως έπρεπε όντω να συζητηθεί το θέμα. Γιατί ορισμένοι διστάζουν λόγω της πολιτικής κατάστασης ή λόγω άλλων ε, δυσκολιών ή επιφυλάξεων. Το θέμα για την Κένια, τη Σομαλία, η επιχείρηση της Σομαλίας. Έχουμε συμφωνία με την Κένια για να βοηθήσουμε ώστε να δικάζονται οι πειρατές που θα συλλάβει η U4 Αταλάντα στην ανοιχτή θάλασσα. Ξέρω πως δεν είστε ικανοποιημένοι, αλλά έχει υπάρξει συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τμήμα της δέσμευσης των κενιατών και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε. Προσπαθούμε να έχουμε τις ίδιες συμφωνίες με τη Σεχέλα στην Τανζανία, ώστε να μπορούν να δικάζονται οι πειρατέ που ίσως συλληφθούν. Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι ξέρω πως η Κομισιόν προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτή την υπόθεση την Κένια για να βελτιώσει τι δυνατότητές τη, διότι ορισμένε από τι χώρε για τι οποίε μιλάμε, η Κένια ίσω λιγότερο από ό,τι άλλε, αλλά ε, έχουν πολύ αδύναμα δικαστικά συστήματα και λιγοστούς πόρους στη διάθεσή τους για να βοηθήσουν σε αυτή την υπόθεση. Και γι' αυτό και έχει νόημα εμείς να τους βοηθήσουμε και η Κομισιόν να δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα. Για την ε, ΚΕΠΑ Προσπαθούμε να βελτιώσουμε συνέχεια την αισθητή, όχι μόνο απλά επειδή υπάρχει, αλλά πιστεύουμε σε αυτήν, πιστεύουμε πως υπάρχει η ζήτηση, πιστεύουμε πως είναι επιτυχής μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω πώς το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να παίξει ρόλο στη Γεωργία. Ούτε στον Άτσε. Εγώ νομίζω πως σε αυτές τις δύο χώρες κάναμε πολύ επιτυχείς παρεμβάσεις, για να σας δώσω μόνο κάποια πρόσφατα παραδείγματα. Θα μπορούσα να πω δύο λόγια παραπάνω στην, για το Αφγανιστόν. Η ESTP είναι η U-POL δηλαδή ε, θα πρέπει να, να συνεχιστεί η αποστολή αυτή και ξέρω τα σχόλιά σας γι' αυτό. Ε, έχει βελτιωθεί απίστευτα από τότε που ξεκίνησε. Έχω μεταβεί εκεί, εδώ έχω δει, έχω δει την ε, μονάδα αυτή σε δράση. Έχω δει τον Υπουργό Εσωτερικών του Αφγανιστάν που μα είπε ότι σε στρατηγικό επίπεδο συνεργάζεται πολύ στενά με αυτή την αποστολή. Θα πρέπει να κάνει περισσότερα επιτόπου, πιθανότατα. Αλλά εκεί ε, προσκρούμε στο θέμα τη ασφάλεια. Είναι δύσκολο. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερε βελτιώσει για την ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ, την ε, ΙΣΑΦ, τη συνεργασία με την Europol ε, θα πρέπει να έχουμε μια πρακτική προσέγγιση. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε να βρεθεί πρώτα η πολιτική λύση. Θα πρέπει να έχουμε πρακτική προσέγγιση λοιπόν προς αυτό. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όταν δηλαδή όσο πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καλωσορίζουμε οποιαδήποτε οργάνωση είναι η e για τις χώρες που θέλουν να συμβάλλουν και που δεν είναι μέλη της Ένωσης. Θα πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτες. Ήδη βασιζόμαστε στην στήριξη της ε, Νορβηγίας, της Τουρκίας, της Αμερικής, ε, του Καναδά. Ένα σωρό χώρες συμβάλλουν, αλλά θα πρέπει καθημερινά να ανοίγουμε στη διαδικασία ώστε και τα κράτη που δεν είναι μέλη να θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν. Ε, τον ίδιο τρόπο η Σουηδία ως ε, χώρα που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ ε, εμείς βάζουμε κόσμο στην ΆΙΣΑΦ και στις σχετικές επιχειρήσεις και ελπίζουμε πως και ο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ μάλλον θα είναι έτοιμο να συμβάλλει σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπως και εμείς. Για το Αφγανιστάν, μεγα πόροι εδώ για όλους τους λόγους που αναφέρετε και για πολλούς άλλους ακόμα. Νομίζω πως κάθε κράτος της Ένωσης συμμετέχει. Είτε θετικά είτε με τη διμερή συνεργασία έχουμε την έννοια του PRT το οποίο διοχετεύει πολλούς σπόρους στο Αφγανιστάν, αλλά ήταν και ένας τρόπος κατακαιρματισμού της συνεργασίας. Εμείς θεωρήσαμε πως η Ένωση μπορεί να παίξει ρόλο όσον αφορά την πιο συντονισμένη προσέγγιση σε αυτό που αποκαλούν οι Αμερικανοί την ε, αναζήτηση των ε, πολιτών, να κάνουμε και εμείς το ίδιο πράγμα, δηλαδή να διοχετεύσουμε τις διμερείς μας, τους διμερείς μας πόρους σε κάποιους βασικούς τομείς, πέρα από τα όσα κάνουμε στο στρατιωτικό τομέα. Αυτή είναι μια από τις βασικές συζητήσεις που έχουμε με την ε, ε, στους Υπουργούς ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, το συζήτησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και προσπαθούμε να εκπονήσουμε ένα βελτιωμένο σχέδιο για την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά έχουμε λοιπόν επιτάπητος για τους πολλούς και διάφορους λόγους που αναφέρθηκαν ήδη κατά τη συζήτηση εδώ. Η υποπτία, η επιτήρηση της θαλάσσης, ναι και εδώ μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία. Πολλά γίνονται για το περιβάλλον, για την αλληλεία, για την ακτοφυλακή. για την ασφάλεια στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Και αν δούμε τη δική μας υπόθεση, τη σουηδική περίπτωση ή τη συνεργασία στην Βαλτική θάλασσα που έχουμε πολιτικά συστήματα και στρατιωτικά συστήματα που λειτουργούν. Υπάρχει χώρος για βελτιώσεις στην συγχρονισμό των δύο συστημάτων και πάλι εξοικονομούνται χρήματα και κάποιες από τις πληροφορίες που έρχονται από την πολιτική παρακολούθηση και παρατήρηση των θαλάσσιων περιοχών ε, στο στρατιωτικό πλαίσιο ή αντιστρόφως ανάλογα. Υπάρχει, γίνεται λοιπόν πολύ οριζόντιο συντονισμό και θα πρέπει να γίνει όλα και περισσότερο μόλι αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό. Να δούμε ακριβώς τι κάνουμε και πού θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερο συντονισμό. Ορισμένα από αυτά που κάνουμε είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα για την περιφερειακή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρεμβαίνει μόνο όταν υπάρχει προστιθέμενη αξία. Πάντως σίγουρα υπάρχει χώρος βελτίωσης. Το Δεκέμβριο ελπίζω πως θα μπορέσω να σας εξηγήσω πόσο και πώς προχωρήσαμε. Τώρα, η κυρία Τζανέλα νομίζω πως θα είναι σε καλύτερη θέση για να μιλήσει για το MPT. Υπάρχει βελτιωμένο διεθνές περιβάλλον να προσπαθήσουμε να έχουμε πρόοδο σε αυτά τα θέματα. Όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση Μπάρακ είναι ε, υπέρ της μη διάδοσης, αλλά και γιατί μπορούμε, υπάρχουν περισσότερα κράτη μάλλον τα οποία ενδιαφέρονται και όπως σας είπα η αναλύση Τζανέλα θα σας δώσει πολύ καλύτερες εξηγήσει για αυτό το περίπλοκο θέμα και το τι συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη, έχουμε ακόμα έξι ε, παρεμβαίνοντας. Σας ζητώ να είστε σύντομοι γιατί έχουμε γεμάτη ημερήσια διάταξη σήμερα. Ο κύριος Κυρίλοφ. Thank you, Ευχαριστώ σύντομα. Κι εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο Φανόρδεν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι και εγώ εκφράζω ανησυχία. Διάβασα πρόσφασα, πρόσφατα για την προσπάθεια αναθεώρησης της κατάστασης και από πλευράς των Αμερικανών. Υπάρχουν δύο σχολές. Η μία είναι να συνεχίσουμε και να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας με μη στρατιωτικές επιχειρήσεις και η άλλη σχολή είναι να γίνει μια πλήρης αναθεώρηση. Με κατάρτιση, με ανοικοδόμηση. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την ιστορία και το παρελθόν της χώρας αυτής. Και οι Βρετανοί μάλιστα πολύ, ακόμα και οι Ρώσοι Νομίζω ότι προσπάθησαν να κάνουν πολλά στο μη στρατιωτικό τομέα, αλλά γενικά μιλώντας, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος εκεί δεν αφήνει, οι Αφγανοί δηλαδή δεν επιτρέπουν ξένη επέμβαση για πολύ εκεί. Ακόμα και αν στην αρχή υπάρχει ενθουσιασμός, οι Ταλιμπάν πώς να το πω, ήταν εχθροί. Έτσι τους έβλεπε ο κόσμος. Τώρα είμαστε όμως σε μια διαφορετική κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να κάνουμε μια μεγαλύτερη διανοητική προσπάθεια. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε να βάλουμε χρήματα σε άλλους τομείς αν συνεχίζουμε με στρατιωτικούς, ακόμα και μη στρατιωτικούς στόχους, φοβάμαι ότι θα μας μισούν περισσότερο. Και όσο περισσότερο μας μισούν, καταλαβαίνετε, είμαστε από άλλο πολιτισμό, από άλλη περιοχή. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Θέλω να αναφερθώ επίσης και στο κοσυφοπέδιο. Κύριε Πρέσβη, πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Την προηγούμενη εβδομάδα πράγματι συζητήσαμε με τον Πίτερ Φιτ σημείωσα ότι είπατε ότι τώρα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε το μέγεθος της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος που υπάρχει και πρέπει να σταματήσει. Αυτό τι σημαίνει. Ότι προσπαθούμε, ότι αγωνιζόμαστε. Με ό,τι έχουμε. Τι έχουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κίνημα πολύ αποφασιστημένο, ναι, αλλά όσο και σου αρέσει όλες, όμως επιτίθεται. Δεν νομίζω ότι οι γκάγκστερς αυτοί, οι παλιωμοδίτικοι, έχουν σύνδεση με τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί βλέπουν ήδη κάποια αποτελέσματα και θα συνεχίσουν να τους, αγων... να... τους πολεμάνε. Είπαμε κάποια στιγμή ότι θέλαμε να δώσουμε ανεξαρτησία στο κοσφοπέδιο. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε. Ακόμα και αν υπήρχαν και άλλες λύσεις, τώρα έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι τα πράγματα μπορεί και να χειροτερέψουν. Ας μην είμαστε δηλαδή πάρα πολύ αισιόδοξοι και τότε θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ας δείτε τι έγινε με Γερμανούς που είπαν ότι οι τρομοκράτες τους κατηγόρησαν. Ας προσέξουμε λοιπόν και να ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα εκεί να είσαστε σύντομοι στα σχόλιά σας. Μη θέτουμε σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του Κωσυφοπαίδειου σήμερα. Ερωτήσεις να κάνετε για να μπορούμε όλοι να κάνουμε ερωτήσεις και να μπορέσουμε να έχουμε πραγματική ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη. Ο κύριος Γουλτιέρη, το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. καθότι η εισήγησή σας ήταν ε, πληρέστατη και συμφωνώ με τη θετική σας κρίση ε, για αυτή την πρώτη δεκαετία της ε, ΚΕΒΑ. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σε μία πτυχή που θεωρώ πως ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί πιο εις βάθος. Ακριβώς επειδή η ΚΕΠΑ μεγαλώνει και ε, φαίνεται να αντιμετωπίζει μια κρίση ενηλικίωσης, ε, ακριβώς ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέσα, μάλλον ποια είναι τα προβλήματα των μέσων συλλογής πληροφοριών, στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού του πολιτικού με το στρατηγικό σχέλος, παρακολούθησης των επιχειρήσεων, ποια είναι τα προβλήματα αυτής της σημερινής δομής της ΚΕΠΑ. Θα ήθελα να έχω μια κρίση του κυρίου Πρέζου για την καταλληλότητα των μέσων που υπάρχουν και για την γνώμη του για το πώς αυτά θα ενισχυθούν. Και κάτι ακόμα, ένα συγκεκριμένο μέσο, δηλαδή ο σημερινός προβληματισμός που υπάρχει για τις απειλές σε θέματα διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Ακριβώς αυτός ο προβληματισμός που πιστεύω πως κατά τη διάρκεια της Σουηδικής ε, Προεδρίας θα πρέπει να ευαθυνθεί. Πώς λοιπόν ε, αυτός ο προβληματισμός θα γίνει με τον κατάλληλο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Merci, Monsieur Ευχαριστούμε, κύριε Ζέμκη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, μας είπατε να είμαστε σύντομοι, γι' αυτό και εγώ θα φροντίσω ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Πρώτο λοιπόν το σχόλιο μου. Είναι καλό το ότι η Σουηδική Προεδρία θέλει να ασχοληθεί με το θέμα των ομάδων μάχης και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Νομίζω ότι είναι τρομερό για την ασφάλεια να παριστάνετε ότι κάνετε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το κάνετε. Οι μικτές ομάδες μάχης ε, πιστεύαμε ότι θα ήταν μάλλον ε, φάνηκε ότι ήταν εικονικές. Πολλές χώρες είχαν επιλέξει να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες μάχης και τελικά τώρα δεν έχουμε καμία τέτοια περίπτωση, δεν έχει αναπτυχθεί καμία τέτοια ομάδα μάχης. Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να αποφασίσουμε θα έχουμε πραγματικές ομάδες μάχης ή θα το ξεχάσουμε. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Απορρέει από την τρέχουσα κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου δουλεύουμε ήδη πάνω στον προπολογισμό του 2010. Όπως πάντα υπάρχουν επιστώσεις υποχρεώσεων για μικτές δράσεις, κοινέ δράσεις στον τομέα της ασφάλειας. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε προβεί σε ανάλυση του σχεδίου προϋπολογισμού και αν ναι, είναι η άποψή σας ως Προεδρία. Και εσείς ως Προεδρία έχετε προτάσεις για το τι θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στον προϋπολογισμό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Μαυρονικόλας έχει το λόγο. Ναι, να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον κύριο Σκόκ για μια λεπτομερή αναφορά σε όλες τις τυχές που αφορούν την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Θα έλεγα ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνονται παγκοσμίω ότι είναι ειρηνικές, αποδοτικές και τοποθετούνται στην πρώτη, σε ένα πρώτο επίπεδο αποτελεσματικότητας με ορθό τρόπο. Ε, στον τομέα των battle groups, των μονάδων ταχείας αντίδρασης, ε, σίγουρα είναι ένας τομέας ο οποίος πρέπει να το ξαναδούμε. Πιστεύω ότι ασχολήθηκαμε για πολλά χρόνια με τα battle groups και η Υπουργή Άμυνας και στο τέλος της ημέρας έχουμε δημιουργήσει ένα υπέρμετρο αριθμών μονάδων ταχείας αντίδρασης που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, που δεν είναι αποτελεσματικές και που πολύ περισσότερο υπάρχει το βέτο της κάθε χώρας για το Battle Group το οποίο συμμετέχει. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της θαλάσσιας επιτήρησης που εγώ πιστεύω ότι η κοινή πολιτική της άμυνας ανοίγονται διάφοροι τομείς όπως είναι η θαλάσσια επιτήρηση όπου οφείλουμε να ενισχύσουμε αυτόν τον τομέα να θέλουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Συμφωνώ απόλυτα με την αρχική σας τοποθέτηση ότι μπορεί να μην έγιναν πολλά είναι όμως βήμα-βήμα και είναι καιρός να προχωρήσουμε έστω ακόμα ένα βήμα με τη νέα Προεδρία. Τελειώνω με την αναφορά ότι για μένα τουλάχιστον η κοινή άμυνα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι πιστεύω όπως θέλω να πιστεύω ότι το νιώθετε κι εσείς ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οικοδομήσουμε και μια κοινή εξωτερική πολιτική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Witt. Thanks very much, uh, President. I've had the advantage of seeing... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είχα το πλεονέκτημα να δω τις αποστολές στην Βοσνία, Ερζεγοβίνη